Καλησπέρα σας. Πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει καμία πρόταση τροποποίησης ή να τη δεχτούμε. Δεύτερον, υπάρχουν εκπρόσωποι από τα κοινοβούλια των χωρών του Περσικού κόλπου που έχουν έρθει εδώ επίσκεψη στην Ένωση. Τους χαιρετίζουμε. Και τώρα το πρώτο θέμα, η ανταλλαγή απόψεων με τον Χωσέ Ράμος και Χόρτα. εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Γουινέα Μπισάου και πρώην πρόεδρος του ε, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου για το Τιμόρ Λέστε και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Θα μας μιλήσει λοιπόν και μετά θα συζητήσουμε. Ορίστε κύριε Χόρτα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω ξαναέρθει και άλλες φορές σε αυτό το κτίριο εδώ και 30 χρόνια πολλές φορές και πάντοτε τύχαινα <clears throat> πολύ καλής υποδοχής και κάθε φορά παρουσίαζα τα του Τιμόρ. Δεν θέλω να φάω πολύ χρόνο από το κύριο θέμα που θα μας απασχολήσει, αλλά ήθελα να πω ότι πριν από μερικές εβδομάδες ήμουν στον Ταβός και συνομιλούσα με μια ομάδα Ευρωπαίων, μερικοί από τους οποίους σχολίαζαν θετικά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στην Ευρώπη. Ένας όμως είπε ποιος ανόητος πρότεινε την Ένωση για το Νόμπελ Ειρήνης και είπα εγώ. Εξεπλάγει πολύ και σε μερικές, πριν από μερικές εβδομάδες στη Λισαβόνα ο πρόεδρος Μπαρόσο αν και η Άννα Γκόμες είναι ταγμένη κατάλληλα τέλος αποσιοποιητικά για την προηγούμενη εβδομάδα στη Λισαβόνα. Γιατί πρότεινα εγώ την Ένωση για το βραβείο Νόμπελ, γιατί μέχρι τώρα η Ένωση ήταν απομονωμένη στον ΟΗΕ και στη Νέα Υόρκη και στη Γενέβη, στην πρώην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μόνη της για να μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τη δημοκρατία και πλήρωνε τίμημα στις διεθνείς της σχέσεις γι' αυτό. Εσείς είχατε αναλάβει την πρωτοβουλία για μερικές από τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες συμφωνίες όπως Λομέ Κοτονού, το Everything But Arms, προσπαθώντας να προωθήσετε δίκαιες εμπορικές σχέσεις με χώρες του τρίτου κόσμου. Και βέβαια καταφέρατε να ξεπεράσετε την τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό καθόμουν εκεί μια μέρα και έγραψα στην Επιτροπή Νόμπελ ένα πολύ μακροσκελές πόνημα όσο και να παραξενεύτηκε κάποιος εκεί στον Ταβός ότι κάποιος από ένα μικρό, από μια μικρή και μακρινή χώρα του κόσμου πρότεινε το Νόμπελ Ειρήνης για την Ευρώπη. Ίσως αν το είχε προτείνει Ευρωπαίος θα θεωρούνταν ύποπτο. Αλλά ένας σχετικά άγνωστος από μία μικρή χώρα που όμως έχει επωφεληθεί από όλα όσα έχετε από όλες σας τις προσπάθειες. Και τώρα γιατί τη Γουινέα Μπισάου όταν μου ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας Μπαν Κιμούν να οριστώ ως ε, ειδικό του εκπρόσωπο στη Γουινέα Μπισάου ή για τη Γουινέα Μπισάου. Είχαμε συμφωνήσει να γίνουν όλα αυτά σε επίπεδο της Γενικής Γραμματείας, όχι χαμηλότερο, και συνάντησα και όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη και πολλοί, πολλούς άλλους το CPLP, το CDAU και όλοι αναγνώρισαν ότι εδώ και πολλά χρόνια η διεθνής κοινότητα δεν είχε ασχοληθεί στα σοβαρά με τη χώρα αυτή. ούτε στις καλές εποχές ούτε στις άσχημες. Στις άσχημες εποχές δεν έκανε καμία προσπάθεια, στις καλές εποχές πάλι αδιαφορούσε. Ο ΙΕ βέβαια είχε πάντα πολύ περιορισμένη παρουσία στη Γουινέα Μπισάου και γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε να θεωρηθεί επίπεδο υπογενικής γραμματείας αυτή η θέση όπως η αποστολή για το Αφγανιστάν ή το Μαλί. Αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας ζήτησε να γίνει μία, να μου να κάνω μία παρουσίαση αξιολόγηση της κατάστασης και να υποβάλω προτάσεις τον Μάιο εάν χρειαστεί δε και να αναδιοργανωθεί η παρουσία του ΟΗΕ στη Γουινέα Μπισάου. Έτσι ώστε να αλλάξουν κάπως τα πράγματα από την διεθνή και σταθερή αυτή αδιαφορία. Διότι όταν δεν υπάρχει σαφής στόχος ούτε τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού τότε φυσικά αποτυχαίνουμε. Και είτε πρόκειται για τον ΟΗΕ είτε για την Ένωση, χάνει αξιοπιστία η διεθνής κοινότητα. Γιατί μετά από 40 χρόνια θα μας πούνε υπάρχει ακόμη τόσο μεγάλη φτώχεια στη Γουινέα Αγγισάου. Εντάξει, φταίνει και η πολιτική της. Αλλά και η διεθνής κοινότητα. Τις προάλλες πήγα σε ένα στρατηγείο στη Γουινέα Μπισάου και σπάραξε η καρδιά μου. Πώς μπορούν άνθρωποι να φέρονται σε άλλους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο. Το στρατόπεδο, το αρχηγείο του στρατού δηλαδή, η κουζίνα, οι κοιτώνες όλα ήταν πολύ άσκημα, σε πολύ άσκημη κατάσταση. Φυσικά αυτά είναι και οι πολιτική και στη Γουινέα Μπισάου και στη χώρα μου. Πρέπει όμως να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Και κυρίως όσοι λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί να μην υπάρχουν αξιοπρεπείς κοιτώνες και κουζίνες στο αρχηγείο του στρατού. Ο τρόπος με τον οποίο φέρονται στους στρατιώτες στη Γουνέα Μπισάου δεν είναι ανθρώπινος. Είπα λοιπόν και στο Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι θα πω την αλήθεια για όποιον θέλει να την ακούσει. Ότι δεν θα περιοριστώ να υπογράψω και να αναφέρω πράγματα και κείμενα που θα τα έχουν γράψει άλλοι για μένα. Η κατάσταση που είναι σήμερα δεν χαρακτηρίζεται από ένοπλη σύραξη, δεν είναι μαλλί, δεν είναι Κονγκό. Υπάρχει βέβαια μεγάλη κρατική ανοργανωσιά, παρέμβαση του στρατού στα πολιτικά, αλλά και οι πολιτικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν καλύτερα, τίποτα καλύτερο. Επομένω, με, καλύτερη διεθνή, με καλύτερο διεθνή συντονισμό ελπίζουμε οι αρχές στη Γουινέα Μπισάου μαζί με μια νόμιμα ελεγμένη κυβέρνηση και κοινοβούλιο να μπορέσουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα που να οδηγήσει στη διοργάνωση εκλογών το Νοέμβριο. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν αυτό περιμένει και η Ένωση και ο ίδιος εγώ αυτό προσδοκώ. Να γίνουν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές προς τα τέλη του έτους. Προτείνω όμως να επανορίσουμε τι εννοούμε με την μετάβαση. Συνήθως μετάβαση νοείται η περίοδος από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Για τη Γουινέα Μπισάου όμως δύο μεταβατικές φάσεις πρέπει να υπάρξουν. Από σήμερα μέχρι τις εκλογές και δεύτερη φάση από τις εκλογές και μετά. Ελπίζοντας βέβαια η κυβέρνηση να είναι σταθερή και να μην αμφισβητηθούν οι εκλογές για να έχουν όλοι το αίσθημα ότι δεν έχει χάσει κανείς. Δηλαδή το πρώτο κόμμα να ζητήσει από το δεύτερο ή τρίτο μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας για μερικά χρόνια. Ξέρω ότι δεν θα γίνει εύκολα αυτό. Θα χρειαστεί κάποιος εξαιρετικός πρωθυπουργός, ένας χαρισματικός ηγέτης για να μπορέσει να κρατήσει ένα συνασπισμό για 3, 4, 5 χρόνια. Και εσείς στην Ευρώπη καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει ένα συνασπισμός, πόσο μάλλον σε χώρες σαν τη Γουινέα Μπισάου. Αλλά είναι μια πρόκληση που τη θέτουμε στους πολιτικούς ηγέτες εκεί. Η δεύτερη αυτή φάση λοιπόν θα την έλεγα ανοικοδόμηση του κράτους αναδόμηση του κράτους. Γιατί σχεδόν όλα πρέπει να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Η πρόκληση για τους πολιτικούς της Γουινέας Μπισάου έγκυται στην αναγνώριση των προβλημάτων της χώρας τους τις τελευταίες δεκαετίες. Τέχονται διεθνή βοήθεια με τρόπο παρεμβατικό, δηλαδή τα Υπουργεία Οικονομικών και άλλα πρέπει να Αναδιοργανωθούν από ξένους διεθνείς εμπειρογνώμονες του Δουνουτού και άλλους. Ελπίζω και η Ένωση που υπήρξε αρκετά γενναιόδορη προς τη Γυναία Μπισάου μέχρι τώρα θα κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Χρειάστηκαν και κυρώσεις βέβαια, ήταν αναπόφευκτο, αλλά κάνατε, πράξατε το σωστό. Δεν ακυρώσατε δηλαδή προγράμματα που ωφελούν τον απλό πολίτη. Θα σας ζητούσα λοιπόν να συνεχίσετε αυτά τα προγράμματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή τις υπηρεσίες της οργανώσεις του ΟΗΕ. Αν θεωρείτε ότι δεν πρέπει ή δεν μπορείτε άμεσα να κάνετε οτιδήποτε. Υπάρχουν εκκλησίες, η ΜΚΟ, ο ΟΗΕ και εγώ και μπορείτε λοιπόν να βρείτε τρόπους να συνεργαστείτε, να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας που να οδηγήσουν στις εκλογές. Τώρα το οργανωμένο έγκλημα και τα ναρικοτικά. Έχουν ακουστεί πολλά στο διεθνή τύπο για το ότι η Γουινέα Μπισάου έχει γίνει χώρα κέντρο διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αφρική. Εγώ διαφωνώ διότι αυτές, αυτά τα συμπεράσματα, αυτές οι αξιολογήσεις δεν με έπεισαν ακόμη και αν προέρχονταν από οργανώσεις του ΟΗΕ ότι η Γουινέα Μπιζάου είναι ναρκοχώρα. Μου είχαν πει πριν να πάω ότι παντού φαίνεται πλούτος δυσεξήγητος. Εγώ δεν είδα πολλές BMW εκεί πέρα, μία-δύο το πολύ. Πήγα και στο σπίτι εκείνου που τον ονόμαζαν βασιλέα των ναρκωτικών στη Γουινέα Μπισάου. Είναι ένα σπίτι μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα. Μου είπαν ότι έχει ψηλούς τείχους γύρω από τον κήπο και δέκα αυτοκίνητα μέσα. Είναι ο αρχηγός του στρατού. Και του είπα μπορώ να επισκεφθώ το σπίτι σου. Μου είπε ναι, την επομένη πήγα. Μένει σε ένα σπίτι που δεν κοστίζει παραπάνω από 10.000 δολάρια για την κατασκευή του. Από λασπότουβλα και λίγο τσιμέντο ούτε ένα δε αυτοκίνητο. Μετά μου είπαν ότι είχε μία πολυτελή βίλα στην Τακάρ, μπροστά στη θάλασσα. Ρώτησα εκεί στην Τακάρ, πού είναι το σπίτι του στρατηγού Ιντάι, μου είπαν δεν ξέρουμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα οργανωμένου εγκλήματος ή ναρκωτικών σε ολόκληρη την Δυτική Αφρική, αλλά τα ναρκωτικά συνεχίζουν να παράγονται στην Νότια Αμερική, Κολομβία, Βολιβία, Περού. Από εκεί θα με πλοίο καταλήγουν στην Αφρική, είτε στη Γουνέα Μπισάου, είτε στο Μαλί, είτε οπουδήποτε αλλού. Transit through Mauritania, Morocco and land in Europe. The epicenter Υπάρχουν δύο επίκεντρα, η Νότια Αμερική και η Ευρώπη. Αν λοιπόν δεν καταργηθεί η παραγωγή των ναρκωτικών, αν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν μέσω της παιδείας ή της αστυνόμευσης να σταματήσουν τη διακίνηση των ναρκωτικών, ή ψέγεται μόνο τους Αφρικανούς, οι οποίοι είναι τα θύματα αυτή τη δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην Νότια Αμερική και την Ευρώπη. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν για να αποτραπεί η κίνηση αυτή των ναρκωτικών προς τη Δυτική Αφρική. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα όσο λέγεται, αλλά είναι αρκετά σοβαρά ώστε να πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα και η Γουινέα Μπισάου είναι τόπος όπου μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αν η Ευρώπη παραμείνει σταθερή, αν μπορέσει να τους βοηθήσει να οργανώσουν μία μικρή μονάδα θαλάσσιας αστυνόμευσης, γιατί μην ξεχνάτε ότι περισσότερη παράκτια αλληλεία εκεί γίνεται από ευρωπαϊκά πλοιάρια, υπάρχει παράνομη αλληλεία από Ευρωπαίους που λόγω τους οποίας χάνει πολλές χιλιάδες δολάρια η Δυτική Αφρική. Υπάρχει και λαθρεμπόριο όπλων. Η Γουνέα Μπισάου όμως θα μπορούσε να γίνει μια όαση ηρεμίας γιατί δεν υπάρχει εκεί εθνοτική βία ούτε ακραίες θρησκευτικέ απόψεις, τρεις θρησκείες εκεί συνυπάρχουν ειρηνικά και θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει υπόδειγμα. Είδα εκπροσώπους των μουσουλμάνων που είναι η πλειοψηφία καθολικών και προτεσταντών. Και οι τρεις αντιπροσωπείες συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτέ, σταματάω εδώ ζητώντας Εάν υπάρχουν κονδύλια που θα δοθούν στη Γουινέα Μπισάου, αν και αυτά όλα έχουν παγώσει λόγω του πραξικοπήματος, παρακαλώ μην τα δώσετε σε άλλες υποθέσεις όπως το Μαλί, που είναι τώρα στην επικαιρότητα, αν δεν μπορείτε να τα χορηγήσετε λόγω της πολιτικής κατάστασης, χορηγήστε τα στον ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ. Εκτός αν δεν έχετε εμπιστοσύνη ούτε σε μένα. Δώστε τα στη UNICEF ή στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής. Σας ευχαριστώ και ο Θεός μαζί σας. I think Πάρα πολύ σαφήν όσο μας είπατε. Και τώρα, ο κύριος Σαλαφράγκα να σας δώσει ένα λάκτισμα για τη συζήτηση, για παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Έχει το λόγο κύριε Σαλαφράγκα, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ράμου Σόρτα. Ακόμη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επανειλημμένως τα έχουμε συζητήσει και ειλικρινά σας ευχόμαστε κάθε τύχη για την ε, υλοποίηση της εντολής σας που σας ανέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το 1974 ξεκίνησε η ιστορία της ανεξάρτητης Βουνίας Μπισάου μετά την ε, ε και δημοκρατισμό, μετά τον εκδημοκρατισμό μάλλον της Πορτογαλίας και είχαμε ε, τον κύριο Βιέρα, τον κύριο Γιάλα, τον πρόεδρο, κατά τη δολοφονία του κύριου το 2009 και τελικά είχαμε το γνωστό πραξικόπημα. Μας τα είπατε πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι η κατάσταση στην Γουινέα Μπισάου δεν είναι ακριβώς η ίδια με την κατάσταση που δηλαδή στο Μαλί. Αλλά βεβαίως και δεν μπορούμε παρά να κάνουμε παραλληλισμούς με τέτοιες ε, χώρες, Μαλί, Μαυρτανία. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το είπε ο ΙΕ που το 2004 είπε ότι είχαμε φοβερές ροές από την Νότια Αμερική που παράγεται κοκαίνη προς τις χώρες του κόλπου της Γουινέας. Βέβαια έχουμε εδώ και την Νιγηρία που και αυτή τη χώρα την χρησιμοποιούν για αυτές τις ροές των ναρκωτικών. Το ίδιο και για την ε, ηρωίνη του Λάος, τη Μιανμάρ, της Κίνας, του Πακιστάν και της Ειρήνης σε διάφορες άλλες χώρες. Προκειμένω για ναρκοχώρα, η οποία τη σήμερα ημέρα ηγείται όσον αφορά την παραγωγή αυτών των ναρκωτικών που μετά εξάγεται στην Ευρώπη. Βεβαίω και άλλο των ναρκωτικών είναι και η χώρα μου, η Ισπανία. Επομένω, όλα αυτά με μεγάλη ειλικρίνεια μα τα είπατε. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Νότιο Ατλαντικό είναι πάρα πολύ βασικό για όλα όσα μα απασχολούν σε σχέση με την παγκόσμια ασφάλεια και έχουμε επίση και τη γεωπολιτική που αγγίζει και το Σαχέλ. Άρα γι' αυτό μα ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα για την οποία μα μιλήσατε. Επίση, να δούμε ότι και στα πλαίσια τη κατοχή των ναρκωτικών, επίση, πρέπει να βοηθήσουμε τι προσπάθειε που καταβάλει ο ΕΕ. Έχουν γίνει δύο φάσεις. Πρώτα-πρώτα ομαλοποίηση και διεξαγωγή εκλογών. Για πέστε μας μήπως είναι δυνατόν να μας δώσετε κάποιες πιο συγκεκριμένες ημερομηνίε σε σχέση με το εσείς. Πότε βλέπετε να γίνονται εκλογές. Επίσης, είναι αφετηρία εκλογέ. δεν είναι το τέρμα, ακριβώ όπω μα τα είπατε. Γιατί είπαμε ότι έτσι θέλουμε να δούμε πώς θα ανασυγκροτηθούν οι κρατικές δομές στη Γουνία Μπισάου. Και γι' αυτό και με ενδιαφέρει τι θα γίνει με τις εκλογές. Πάντως εκτός από αυτό που μας είπατε για τον στρατιωτικό ε, που είχε ένα σπίτι 10.000 δολαρίων, εσείς τι λέτε για αυτές όλες τις ε, φήμες και ιστορίες, για το ότι δηλαδή όλα τα φορτία ναρκωτικών περνάνε από τη χώρα αυτή. Πώς τα βλέπετε επομένω σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε και πώς θα μπορούσε πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τη χώρα εκείνη. Και φυσικά να ενεργήσουμε σε συνέχεια των όσων θα αποφασίσει ή και έχει αποφασίσει ο ΙΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μας το να μπορούμε να σας ξαναδούμε σήμερα κοντά μας και είναι πολύ ενθρεντικό το ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, εμπειρία διεθνούς πολιτικής. Τώρα εργάζεστε για τον ΟΗΕ, για στην υπηρεσία ε, που ασχολείται με την Γουινέα Μπισάου. Και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ε, Μοιάζουν με τις ερωτήσεις που ήδη υπέβαλε ο συνάδελφος ε, κύριος Σαλαφράνκα. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λιγάκι καλύτερα την γεωπολιτική κατάσταση. Τι ακριβώς διαδραματίζεται στη χώρα αυτή. Γνωρίζουμε ότι ε, αυτή τη στιγμή μένεται πόλεμος ε, εξουσίας ε, ανάμεσα στις διάφορες αφρικανικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να κυριαρχήσουν και σε αυτή τη χώρα. Παραδείγματος χάρη η διαμάχη μεταξύ Αγγόλας ε, και Νιγηρίας αλλά και η Σενεγάλη έχει άμεσα ε, συμφέροντα στην Γουινέα Μπισάου γιατί στη Γουινέα Μπισάου ε, και μάλιστα και συγκεκριμένα σε μια περιοχή που δεν έχει ακόμα οριστεί επακριβώς υπάρχουν πετρελαϊκά κοιτάσματα. Εφόσον μιλάμε για την ε, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών σε όλη αυτή την περιοχή της ε, Δυτικής Αφρικής, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ε, τρομοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο φτάνει και μέχρι την ανοιχτή θάλασσα με την πειρατεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα όλη αυτή την περιοχή. Και επίση ε, θα ήθελα να γνωρίζω Υπήρξε μία πρώτη και ε, κατόπιν μία δεύτερη φάση μετά τις ε, εκλογές. η χώρα αυτή που είναι συνομιλητής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθότι έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού θα μπορούσε στη χώρα αυτή να υπάρξει και να επικρατήσει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και τέλος ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στην χρηματοδότηση αναφερθήκατε στην αποστολή που επιθυμείτε να αναλάβετε. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω η κυρία Άστον και ο κύριος Πίμπαλτς έχουν έρθει σε επαφή με την χώρα αυτή μετά το πάγωμα των κοντιλίων τα οποία προβλεπόντουσαν για τη χώρα αυτή. Αυτά θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του έτους. Ενδέχεται ε, μετά να ε, ξεπαγώσουν τα κονδύλια και ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξεπάγωμα των κονδυλίων να το συνδυάσει με, τις, ε, με τη δική της την υπηρεσία που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ήμουν μία εξ όλων αυτών οι οποίοι αντιστάθηκαν στο να ακυρωθεί η αποστολή στη χώρα αυτή. Εγώ είπα ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ε, στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται μόνο για κάποιους τομείς που υποφέρουν, αλλά γενικότερα υπάρχει πρόβλημα στη Γουινέα Μπουισάου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαφόρων μορφών αποστολές ε, έτσι ώστε να βοηθηθεί η χώρα να ε, ανασυσταθεί και είναι μια χώρα, θα ήθελα να σας και να μην το ξεχνάμε, η οποία είναι μέλος των ΑΚΕ. Εγώ θα ήθελα να περάσω στα αγγλικά. Ε, όταν ήμουν παιδί πρέπει να σας πω ότι ε, μάζευα γραμματόσημα και όταν έκανα την πρώτη μου ομιλία την Παρθενική εδώ ε, στο Κοινοβούλιο ήταν για το Ανατολικό Τιμόρ και τότε για πρώτη φορά προσέκρουσα στο δικό σας το όνομα, ε, κυρίως όταν η χώρα σας ήταν υποκατοχή. Και πρόσφατα μάλιστα ε, ενεπλάκην σε μια έκθεση για το σύνολο της Αφρικής. Λέτε λοιπόν ότι η Γουνέα Μπισάου ε, δεν είναι χώρα με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά σίγουρα είναι χώρα με πάρα πολλά προβλήματα. Ο εισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το Σαχέλ, έχει αναφερθεί στη χώρα αυτή και εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας ε, αυτοκινητόδρομος ε, ή υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος ή μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς που διακινούν ναρκωτικά ε, μέχρι και την Ιγυρία. Σήμερα μας είπατε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι στην Γουνέα Μπισάου είναι μουσουλμάνοι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καθολικοί λόγω της κατοχής των Πορτογάλων. Από το Σιχέλ πάμε στη Σομαλία, στο Αλσαμπά. Ε, και στην πειρατεία. Ε, εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, σχέσεις ανάμεσα στα ναρκωτικά, τους Ισλαμιστές, το λατρεμπόριο ή μήπως όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, είναι μύθοι. Και κάτι άλλο, εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών, εσείς ως πρώην επικεφαλής κράτους, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα των ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι η αποποινικοποίησή τους θα έλυνε το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φέιλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα Να σας ευχαριστούμε που ήρθατε ξανά. Είναι τιμή για μας να παρίσταστε στις συναντήσεις μας. Πρέπει να σας πω ότι εμείς υπολογίζουμε πάρα πολύ τη δική σας ε, εμπειρία και την αφοσιβότητα που έχετε για να φέρετε σπέρα σε αυτήν τόσο δύσκολη αποστολή. Τον Ιούνιο του 2012 εγκρίναμε ένα ψήφισμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε και είχαμε την ε, Άννα Γκόμες, που πρωτοπόρησε και δούλεψε πολύ, ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει με την Βουίνια Μπισάου. Τώρα, αν κανείς έτσι γενικά θέλει να δώσει μια εικόνα της χώρας, σε σχέση με την κατάσταση και πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με τους ε, εκτοπισμένους, τους πρόσφυγες. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι μπορείτε εσείς να μας πείτε. Τι γίνεται και από πλευράς ανθρωπιστικών αναγκών και κινδύνων για τον κόσμο. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Τι ρόλο νομίζετε ότι μπορούμε να λάβουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανασυγκρότηση της χώρας και του κράτους της Γουινέας Μπισάου. ότι πρόβλημα υπάρχει με τους, ε, με, με, τους πόρους από την Ευρώπη, την ε, αναστολή των ε, χρηματικών ροών. Οπότε, αυτά τα, αυτή αυτά τα κεφάλαια τα οποία είχαν διατεθεί για τη χώρα, δεν θα μπορέσει να τα πάρουν οι κάτοικοι της χώρας, αλλά θα χρησιμοποιηθούν τελικά για να συγκρότησε της χώρας. Σε αφορά τις εκλογές. Είμαστε στη μία πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, τεχνικά, υλικοτεχνικά και έτσι δεν γίνεται τώρα να διεξαχθούν οι εκλογές. Πάντως αν μπορείτε, πέστε μας κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί θέλω να γνωρίζω. Εάν θα μπορούσατε να κάνετε έναν υπολογισμό. Πότε δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς εκλογές. Τι ρόλο επίσης μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κατάρτιση προσωπικού για τις εκλογές. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Λέει ο κύριος Μηγές. Ευχαριστούμε για για τη χώρα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο δεύτερο σημείο όπως ε, τα είπατε. Θέλω να μου πείτε κάτι για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αναφέρθηκαν σε αυτό και άλλοι συναδελφοί και πριν από λίγες μέρες ακόμα και χθε. συζητούσαμε για το, την, τη σχέση της χώρας με το εμπόριο ναρκωτικών. Είναι σταυροδρόμι, είπαμε, στη Δυτική Ευρώπη για την κοκαίνη που έρχεται από την Νότια Αμερική. Θα πρέπει βέβαια να μην υπερβάλλουμε, θα πρέπει να βρούμε σωστέ του τους διαστάσεις, αλλά πάντως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον ρόλο της χώρας ως σταυροδρόμιο για την κοκαίνη. Έχω μια έκθεση και τώρα την ε, ολοκληρώνω όσον αφορά τις ε, διατλαντικές μας σχέσεις και τις σχέσεις ε, με Λατινική Αμερική, ΗΠΑ και την δυτική ακτή της Αφρικής. Πάντω θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα σχέδιο δράσης, το ΕΚΟΒΑΣ, που αφορά τα ναρκωτικά. Έχουμε το ΒΟΑΞΙ που αφορά την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τη Δυτική Αφρική. Εμείς το ΚΟΒΑΣ το στηρίξαμε και έχουμε επίσης και την υπηρεσία των, του ΟΗΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε και αυτοί όλοι οι φορείς συνεργάζονται για την κατολέμηση των ναρκωτικών και του εμπορίου εκεί, σε αυτή την περιοχή. Αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτά όλα τα αρχικά, είναι πρόσφατα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει θέμα στην Δυτική Αφρική. άσχετα από το αν η Γουνία Μπισάου είναι το, το, το χειρότερο ναρκοκράτος, πάντως υπάρχει θέμα. Είναι ναρκοκράτος. Και φοβάμαι ότι σε όλη την περιοχή της Δυτική Αφρικής τελικά το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η κατανόηση ναρκωτικών, αλλά ότι η χώρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμπόριο ναρκωτικών. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Κύριε Όρτα, έχει το λόγο. Ράμος Κοιτάξτε, ε, θα μπορούσα να απαντήσω σε διάφορες γλώσσες, στα αγγλικά και στα ισπανικά, αλλά περνώντας από τη μια γλώσσα στην άλλη, ενδεχομένως να τα μπέρδευα. Γι' αυτό λοιπόν θα με συγχωρέσετε, ε, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ημερομηνία εκλογών, υπήρξε πρόσφατα στην ακτή του Ελεφαντοστούν μια συνάντηση των ε, εκπροσώπων της Γουνέα Μπισάου και όσον αφορά τις ε, εκλογές προβλέπουν ότι οι εκλογές θα γίνουν φέτος ε, κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Μετά λοιπόν από την, από την επιστροφή μου, όταν επιστρέψω στη Γουνέα Μπισάου, προτίθεμαι να ε, κάνω κάποιες ε, συναντήσεις με εκπροσώπους της, ε, του Αφρικανικού Συνδέσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεμονωμένα σε διμερές επίπεδο με διάφορα κράτη να δούμε τι ακριβώς θα γίνει γιατί τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να ενισχύουν τις περιφερειακές οργανώσεις. Κατά καιρού ε, μπορεί να διαφωνούμε όσον αφορά τη στρατηγική, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα η πολιτική του Γενικού Γραμματέα εδώ και πολλά χρόνια είναι να προσφέρει υποστήριξη σε περιφερειακές οργανώσεις που αντιμετωπίζουν περιφερειακές προκλήσεις. Έτσι λοιπόν ε, θα συνεργαστούμε με την ECOWAS ε, για να δούμε το πλαίσιο λιγάκι ε, το οποίο έχουν συμφωνήσει για την Γουνέα Μπισάου. Και κατόπιν θα συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο της Γουνέα Μπισάου την ακριβή ημερομηνία των εκλογών. Όπως σας είπα λοιπόν προηγουμένως, ελπίζουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου η κυβέρνηση και το νόμιμο κοινοβούλιο, γιατί το κοινοβούλιο δεν έχει ακόμα διαλυθεί, θα παρουσιάσουν ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι τις εκλογές. Και το Μάιο θα παρουσιαστεί ένα ευρύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτά όσον αφορά τις εκλογές. Επ' αυτού, νομίζω το έχω ήδη πει στους αδελφούς και τις αδελφές ε, στη Γουνέα Μπισάου, το έχω ήδη λοιπόν πει ότι επειδή υπάρχουν, ε, υπάρχει καχυποψία ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, ε, στους πολιτικούς ε, ηγέτες και πολλές φορές αμφισβητούν το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρούν ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες προβαίνουν σε ελαφροχειρίες, είναι καλύτερα η Αφρικανική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουν όλη αυτή τη διαδικασία των εκλογών. Σας είπα ότι η εκλογική νομοθεσία έχει συνταχθεί από την Εθνική Συνέλευση. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία της ψήφου. Αλλά ε, την όλη διαδικασία, την οργάνωση, μπορεί κανείς ε, να την αθέσει κάποιον εξωτερικό φορέα, αν δεν μπορεί ότι να το οργανώσει. Και ε, λαμβανωμένων υπόψη ε, των συνθηκών που επικρατούν στη Γουνέα Μπισάου, καλύτερα είναι να τεθεί η διαδικασία της οργάνωσης σε κάποιον εξωτερικό φορέα. Ε, τελικά μπορεί να συμφωνηθεί ότι είναι καλύτερα για τα επόμενα 5-6 χρόνια ε, όπου δεν θα υπάρχει κανένας ηττημένος, θα συμμετέχουν όλοι στην ε, ανασύσταση ε, της χώρας, στην οικοδόμησή της και έτσι αυτό θα οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα την αναδιοργάνωση του στρατού, πρέπει να σας πω ότι συναντήθηκα με το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσία και τους μίλησα για την ανάγκη που αισθάνονται όλοι ε, να αναδιοργανωθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Κατά το παρελθόν, ε, πολλοί ε, έκαναν λόγο για τη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Εγώ δεν θέλω να μιλάω για μεταρρύθμιση, προτιμώ να μιλάω για εξυγχρονισμό. Και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε εκ των έσω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους μίλησα, αυτοί είναι οι ιδρυτές, είναι οι πατέρες ε, της ανεξαρτησίας της Γουνέα Μπισάου. Είναι στα 50 τους, 60 τους και όταν τους βλέπει κανείς αυτή ουσιαστικά είναι η ιστορία της χώρας και δεν μπορούμε λοιπόν να τους ε, αφαιρέσουμε την ευθύνη να σκέπτονται ε, το μέλλον των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα. Ε, θα έρθουν λοιπόν να με βρουν, ε, θα παρουσιάσουν το όρομά τους, ε, μια αναλυτική κατάσταση των προκλήσεων, προκλήσεις ασφαλείας και άλλου είδους και μετά βεβαίως όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Αυτό όμως δεν αρκεί. Θα πρέπει όλα αυτά να τα εξισορροπήσουμε και με τις δυνατότητες που έχει η χώρα. Μπορεί να έχουμε ανάγκες, αλλά δεν μπορούμε να τις καλύψουμε. Και όταν έχει κανείς ε, ε, κονδύλια, πάλι ε, εκ νέου είναι αναγκασμένο να καταφύγει στο εξωτερικό, να αναζητήσει άλλες δυνατότητες για να αντιμετωπίσει αυτές τις αντισυμβατικές προκλήσεις ασφαλείας. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής ότι πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να εξυγχρονίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Γουνέα Μπισάου. Δεν σημαίνει ότι αυτό προηγείται όλων των άλλων προβλημάτων. Όλα επίγουν στη χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ήδη μία μελέτη, έχει ε, παρακολουθήσει για δύο χρόνια ε, τις ένοπλες δυνάμεις ε, ε, η Αγκόλα το έχει κάνει επίσης. Ε, φτάνουν λοιπόν οι μελέτες. Θα δούμε ποιες ε, είναι οι συστάσεις αυτών των εκθέσεων και θα βοηθήσουμε τα στελέχη του Γουινέα Μπισάου για να καταθέσουν ένα σωστό πρόγραμμα βοήθειας της χώρας. Όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να διοργανωθεί το σύνολο του κράτους, ε, όχι μόνο ο στρατός, αλλά και πάρα πολλά άλλα. Όσον αφορά τώρα τα ναρκωτικά και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών στο σύνολο της ε, Δυτικής Αφρικής και η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει γιατί όλα αυτά αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας τρόπος ε, για να το κάνει κανείς είναι ε, να γίνονται καλύτερες ε, έρευνες σε όλη αυτή την ακτή γιατί ακόμα και η Σενεγάλη έχει ένα σύστημα ραντάρ το οποίο όμως φτάνει μόνο μέχρι το αεροδρόμιο. Ό,τι έρχεται από τη θάλασσα η Σενεγάλη δεν μπορεί να το εντεπίσει. Πόσο μάλλον η Γουινέα Μπισάου. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ραντάρ που να εντοπίζει σκάφη ή ε, αεροσκάφη που πλησιάζουν στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει αμελητή, χωρίς καθυστέρηση, μέχρι να οργανώσουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις να υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία ναυτική ασφάλεια. και εδώ χρειαζόμαστε ε, τη βοήθεια της ε, Ευρώπης. Μπορεί να υπάρξει μια πλωτή βάση, ένας πλωτός ναύσταθμος πέρα από τα, από τα χερσαία εδάφη. Εκεί μπορεί να γίνει και η εκπαίδευση, η αποκατάσταση των υποδομών και έτσι λοιπόν θα γίνεται η παρακολούθηση ε, στον αέρα και στη θάλασσα. Και με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί, μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τη διείσδυση ναρκωτικών στη Γουνέα Μπισάου και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορώ να σχολιάσω τα διάφορα συμφέροντα που έχουν οι χώρες ε, στην Γουνέα Μπισάου. Ίσως όταν ε, εκπνεύσει η εντολή μου, ε, αυτό που κάνω τώρα, τότε θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και στις χώρες ΑΠΚΕ ε, δεν υπάρχει ομοφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Γουινέα Μπισάου. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στην ΕΚΟΓΑΣ και την Αφρικανική Ένωση. Είναι νομίζω φυσιολογικό το ότι όσον αφορά τις ε, χώρες ΕΚΟΓΑΣ, ε, την οικονομική κοινότητα Δυτικής Αφρικής, εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους ε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας μονομένα συμφέροντα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ε, τους ε, έχω πει τη γνώμη μας. Η Γουνέμπισά δεν είναι μάλι. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα της όπως ο μάλλον ε, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του Μαλή στη Γουνέα Μπισάου. Ε, δεν ε, έχουμε εμφύλιο πόλεμο και κατ' ουσίαν ποτέ δεν υπήρχε στρατιωτική κυβέρνηση. Ε, εντάξει παρεμβαίνουν, προσπαθούν να επηράσουν, αλλά ποτέ δεν σχημάτισαν κυβέρνηση. Ακόμα και η τρέχουσα κυβέρνηση προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτούς που τους έφεραν βέβαια στην εξουσία. Ο πρόεδρος δεν ήθελε να αναλάβει το αξίωμά του. Είναι ε, μέλος του πολιτικού γραφείου του PHC. Δεν είναι αλήθεια, δεν ισχύει ότι οι στερεωτικοί απέχουν πλήρως, αλλά όπως είπα υπάρχει μια απόσταση. Όσον αφορά τώρα την αποποινικοποίηση ή όχι των ναρκωτικών, Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ένα θέμα ε, το οποίο έχω μελετήσει εγώ. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα ήθελα να τολμήσω να απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Τώρα, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, πράγματι υπάρχει ακραία φτώχεια, ακραία κακή διατροφή, ε, δεν υπάρχει καθαρό νερό. Ακόμα δεν υπάρχει πολιτική ρύθμιση που να είναι αποδεκτή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας παρακαλέσω να επεκτείνετε τη βοήθεια μέσω του γραφείου μου, μέσω της UNICEF, ε, το World Food Program και άλλους οργανισμούς των Αμερικανών. Γιατί οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν κάποια παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες για το προσωπικό που ζει ε, στη χώρα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ενισχύσετε τη χώρα αυτή. Αν δεν μπορείτε να ενισχύσετε άμεσα την κυβέρνηση, τότε ίσως ε, να βοηθήσετε τους ε, ε, οργανισμούς των ΗΕ και της ΜΚΟ. Νομίζω λοιπόν ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν δεν μπόρεσα να απαντήσω σε κάποιες εξ αυτών, ίσως δεν ξέρω, μπορείτε να επανέλθετε. Παρακαλώ. Well, Thank you very much. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χρήσιμη ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ευκαιρία για μας να έχουμε από πρώτο χέρι πληροφορίες για την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και απαντήσατε τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστούμε κύριε Χόρτα. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο.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 right. So we have two votes. Τώρα θα ψηφίσουμε. Πρώτο θέμα, η γνωμοδότηση για τα δικαιώματα των γυναικών στις ε, βαλκανικές υποψήφιες χώρες. Έτοιμοι. Προπολογία 1 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ένα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Okay. Uh, number five. Amen. Πέντε υπέρ κατά εποχές εγκρινείται έξι υπέρ κατά εσ, εγκρινείται συμβιβαστική δύο υπέρ κατά εσ, εγκρινείται οχτώ τροπολογία οχτώ υπέρ Α, κατά είπα. Απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 11 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χες ρίπτεται 13 υπέρ κατά χες γίνεται. 14 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 15 σε 7 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά χες γίνεται, δεύτερο υπέρ κατά χες γίνεται τρίτο υπέρ κατά χες γίνεται τέταρτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έβδομο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαοχτώ, υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Είκοσι, υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται Μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε και την 16 αφού απορρίψαμε τη 14 λοιπόν. Η 16 υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 σε δύο τμήματα πρώτον Α, όχι. Ο 24 μου λένε, 24. 24 με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. εποχέ. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο ηλεκτρονικά Δύο χωρίς κάρτα. Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Ψηφίζουν πάντως υπέρ. Μάλιστα, μάλιστα. 29 λοιπόν υπέρ με τους δύο πρόσθετους. Συγχαρητήρια, εγκρίνεται. Τώρα... Η δεύτερη ψηφοφορία. Συμφωνία Ένωσης Κίνας. Είναι μόνο το σύνολο ηλεκτρονικά. Δύο είπαμε δεν έχουν κάρτες. Λοιπόν, έλξε η ψηφοφορία, έλξε 28 με τους δύο υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ, εγκρίνεται. Κύριε Τάνο, συγχαρητήρια. Τήρια τώρα. τώρα. Okay. Λοιπόν, η κυρία Μαρίσα Ματίας λείπει. Λείπει, απουσιάζει. Α, έρχεται όμως, έρχεται. Να την περιμένουμε λοιπόν κανένα δύο λεπτά μέχρι να προσέλθει. Ε, ναι, Πρέπει να σας πω ότι λόγω της επιτάχυνσης της ημερήσιας διάταξης η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ρούπερτ Τζόι μόλις διορισμένο επικεφαλής της αποστολής μας στο Μαρόκο θα αρχίσει στας 5 αντί 5.30. 5. Θα περιμένουμε ακόμη την κυρία Μαρίσα. Okay. So. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι η πληροφόρηση της κυρίας Ματίας για την ενδέκατη διακοινοβουλευτική συνάντηση Ένωσης Λιβάνου που έγινε στο Λίβανο το Φεβρουάριο. Η δε κυρία Μαρίσα Ματίας είναι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασράκ. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της επίπτωσης της Συριακής κρίσης στο Λίβανο και η αναθεώρηση του εκλογικού νόμου εκεί. Έχει 5-10 λεπτά για να μας τα πει και αυτά και άλλα. Έχει το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ και συμπαθάτε με διότι άργησα. Δεν ήξερα ότι θα αρχίσουμε. Νομίζω αρχίζουμε στις και μισή. Ναι, για να σας πω λοιπόν τι έγινε με την αντιπροσωπεία. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα βασικά θέματα που αφορούν την, ε, Τι, τι, τι, τι, Μιλάμε για τις 15 Φεβρουαρίου πήγαμε και είχαμε επίση την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και διάφορους υπουργού, τον Υπουργό Εξωτερικών, των Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Επίση του επικεφαλεί των πολιτικών κομμάτων, καθώ και κόμματα τη Επιτροπή για Εξωτερικέ Υποθέσει και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίση και τον επικεφαλής του στρατού. Επίσης, με εκπροσώπους διαφόρων μη κυβερνών οργανώσεων που κυρίως έχουν ασχοληθεί με τους πρόσφυγες που έχουν από την Συρία και άλλους παράγοντε και με του οποίου ζητήσαμε μετά τι εκλογικέ μεταρρύθμισης. Θα ήθελα τώρα να δούμε σε τι πλαίσιο κινηθήκε η αντιπροσωπεία. Καταρχήν, είχε καταστεί σαφές ότι η ατμόσφαιρα, το κλίμα ήταν φιλικό ε, κλίμα φύτας ειλικρινίας. Και είχαμε επίσης την πεποίθηση ότι όλοι με τους οποίους είχαμε σε επαφή συμφώνησαν όλοι ότι πρόκειται για την πρόθεση να υπάρχει σταθερότητα ε, και κοινή βούληση όλων των εμπλεκομένων ούτως ώστε να προχωρήσουν προς μια εθνική ενότητα στη χώρα. Βέβαια είχαμε την κατάσταση στη Συρία και όπως γνωρίζετε απεφάσισαν σχετικά οι αρχές του Λιβάνου να αποστασιοποιηθούν από όσα γίνονται στην Συρία. Βέβαια, τα κόμματα και η χώρα έχουν διχαστεί από αυτού. Είναι πολύ αποσχιστική αυτή η προσπάθεια, αλλά τελικά ε, θεωρήθηκε από όλους ότι βασικό είναι να, να η ενότητα της χώρας. Αυτό είναι το πολιτικό κλίμα σήμερα στο Λίβανο. Τώρα, Έχω δύο θέματα τα οποία και εσείς τα αναφέρατε στην εισήγησή σας. Δηλαδή, βασικά το τι θα γίνει, πού θα καταλήξει η κατάσταση στη Συρία, όπως γνωρίζετε. Ο Λίβανος είναι η μόνη χώρα που θα καταληξει η κατασταση της συρια οπως γνωριζετε ο λιβανος ειναι η μονη χωρα που εχει τα σύνορα ανοιχτά, εντελώς ανοιχτά για τους πρόσφυγες. Επομένως, Έχουμε 280.000 πρόσφυγες που έχουμε ανασυρεύσει. Κατά μέσο 3.000 πρόσφυγες έρχονται στο Λίβανο κάθε μέρα. Και επομένως έχουμε εδώ πολύ σοβαρές ε, δυσκολίες. Ε, είναι και το θέμα υλικών πόρων, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του πώς αυτή η ανθρωπιστική κρίση θα τη διαχειριστούν ούτε θεωρούμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση τους επόμενους ε, μήνες, τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι έχει η κατάσταση σε σχέση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όλους όσους ήλθαν στις συναντήσεις. Όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για θέμα που να αποσχολήσει τη διεθνή κοινότητα. Θα πρέπει να μπει στο τραπέζι όλοι πολύ προσεκτικά να το εξετάσουν και εμείς θα πρέπει με την ε, ε, σειρά μας να στηρίξουμε τον Λίβανο, γιατί ακόμα και με την ανθρωπιστική βοήθεια που προβλέπεται είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το εκλογικό νόμο, πολύ σημαντικό είναι αυτό και πρέπει να το συζητήσουμε. Να έχουμε ρώτα απαντήσεις, να το συζητήσουμε όσο είναι πιο ανοιχτά, ότι αυτό το συζητήσαμε και διότι Έχω μια σειρά προτάσεων από της τραπέζες. Τον Ιούνιο αναμένεται να γίνουν εκλογές. Για τον εκλογικό νόμο. Mm. Το κοινοβούλιο δεν συνδυάζει όπως ε, όφιλε, αλλά υπάρχει μια υποεπιτροπή του κοινοβουλίου η οποία μελετά το θέμα και έχουν εντολή να ασχολούνται με αυτό ως ε, ότου κάπου καταλήξει αυτή όλη η ζήμωση. Οπότε συζητούν πρώτον το θέμα το αναλογικό αλλά και το πλειοψηφικό ως συστήματα. Δέκα δε ημέρες αφού πήγαμε εμείς έγινε μια ψηφοφορία στην ειδική αυτή επιτροπή οπότε η κυβέρνηση το κόμμα κατά επίσης ψήφισαν υπέρ της αναλογικής. Να σαν σύστημα ή αναλογική. Επομένως, ακόμα το θέμα ανοιχτό. Πάντως γίνανε αυτές τις ψηφοφορίες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε επόμενες ημέρες και εβδομάδες και να δούμε μήπως θα γίνουν τελικά οι εκλογές όπως έχουν προγραμματιστεί. Δηλαδή τον ε, Ιούνιο. Πέραν αυτών θα πρέπει να σας πω δύο λίγων κάποια άλλα συζητήματα τα οποία συζητήθηκαν όσοι ήμασταν εκεί τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, εκπροσωπήσή τους στον ε, πολιτικό βίο, όλα αυτά τα συζητήσαμε σε μια σειρά από τις συναντήσεις μας. Επίσης συζητήθηκαν και για τη δικαιοσύνη και ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά όσον αφορά τα κυρίως ζητήματα που έχουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι βέβαια ότι θέλετε να το συζητήσουμε τώρα. Thank you very much. Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κυρίλοφ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, γυναικεία δικαιώματα, ο δικαστικός τομέας κτλ. Ένα όμως θέμα ιδιαίτερα είναι καυτό και θα ήθελα να ξέρω αν το συζητήσατε στην επίσκεψη Μετά τα γεγονότα του τελευταίου καλοκαιριού στον πύργο, στον Μπουργκάς, πριν από μερικές εβδομάδες, μετά τις πρώτα από έρευνες δηλαδή, η κυβέρνησή μας σε συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες παγκόσμια και μυστικές θεώρησε ότι μπορεί να πρόκειται για τρομοκρατικό δίκτυο γιατί εδώ υπήρξε επίθεση κατά ολόκληρου λεωφορείου. Και αυτό θέτει ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ένωση γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τρομοκρατικό δίκτυο και άρα πιέζεται η Ένωση να κάνει κάτι. Αυτό το συζητήσατε και ποια είναι η εντύπωσή σας. Διότι όπως σας είπα είναι σοβαρό το πράγμα, πολύ πλόκο, λόγω και της κατάστασης στο Λίβανο και τη Συρία, αλλά πρέπει να το πούμε, αν όχι στην δική σας έκθεση, τουλάχιστον εδώ μεταξύ μας. Μάγιο Νταβίτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε για το Λίβανο, για τη Μέση Ανατολή. Και κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία προηγουμένως ε, πριν από την ψηφοφορία να πείτε ότι σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας μέλη της ε, Γραμματείας ε, Κοινοβουλίων GCC. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρίζα για την έκθεσή της ε, και πρέπει να πω ότι οι εκθέσεις που ακούσαμε, όλα αυτά που μας είπε ήταν ε, πολύ χρήσιμες. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα στοιχεία που μας ανησυχούν. Ε, το ένα είναι ότι οι πρόσφυγες που έρχονται από την Συρία εισβάλλουν σε αυτή τη χώρα γιατί... Αυτοί αντιμετωπίζονται δυστυχώς ως απλοί πρόσφυγες, ε, όχι ως πρόσφυγες πολέμου. Ε, αυτοί λοιπόν καταφεύγουν κυρίως σε γνωστούς και οικογένειες, ε, τεράστιο το βάρος. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους ε, βοηθήσει και να συνδράμει έτσι ώστε και οι αρμόδιες αρχές να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Βεβαίως το βασικό πρόβλημα είναι και νομίζω εδώ η συνάδελφό μας έριξε ένα θέμα, ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί ε, πρέπει να ζητήσουμε από την Βαρόνια Άστον να έρθει να μας πει ποια είναι η δική της η θέση. Γιατί ε, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί ε, επανειλημμένα σε Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Και αν θέλετε να σας πω εγώ τη δική μου τη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς ακόμα και αν Όλα δείχνουν τη Χεσμολά. Το θέμα είναι ότι η Χεσμολά εκπροσωπείται στον κυβερνητικό συνασπισμό ε, μιας χώρας με την οποία έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ε, θα πρέπει να το δούμε και πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις ε, έτσι ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε και τις δικές μας τις απόψεις. Ε, πρέπει να σα πω, είναι λίγο περίεργο το ότι ο επικεφαλής ε, ενός πολιτικού κόμματος ή μιας οικογένειας αν θέλετε επενείται και προβάλλεται στην ιστοσελίδα της Χεσμπολά. Σοσιαλιστές, αναφέρομαι στο σοσιαλιστή. Ε, θα το πούμε πάντως αυτό όταν ε, θα επανέλθουμε. Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο επανέφερε η Μαρίζα. Πρόκειται για το μελλοντικό εκλογικό νόμο. Όπως ξέρετε λοιπόν, ανεξάρτητα από το σύστημα που θα ε, χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, βάσει του συντάγματος οι χριστιανοί προτείνουν τον πρόεδρο, ο πρωθυπουργό έρχεται από τους Σουνίτες, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου έρχεται από τη Χεσμολά και το θέμα όμως είναι ότι την έχει αλλάξει η δημογραφική σύνθεση της χώρας. Ξέρουμε ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις γιατί έχει αλλάξει ε, το δημογραφικό σκηνικό από τότε που βρήθηκε το Σύνταγμα. Γι' αυτό λοιπόν το ένα είναι βέβαια οι δημοκρατικές αξίες που επιθυμούμε να προβάλλουμε, το άλλο θέμα είναι τι υπάρχει σήμερα στο Σύνταγμα. Πιστεύω λοιπόν ένα άλλο θέμα το οποίο δυστυχώς σχεδόν ξεχάστηκε με την πάροδο του χρόνου, είναι σχεδόν ανύπαρκτη συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει ξεχάσει και η διεθνής κοινότητα. Ε, πρόκειται για τη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές του Λιβάνου και το διεθνώς ε, λιβανικό ε, και το διεθνώς δικαστήριο για την περίπτωση Αρίρη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί ναι. για όλα αυτά ε, όσα διαδραματίζονται σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Η κυρία Ντεκάιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να με συγχωρήσει η Μαρίζα γιατί δεν ήρθα την ώρα που έκανε την εισήγησή της. Και εγώ νόμιζα θα ξεκινήσουμε στις 4.30. Οπότε ευνηδιάστηκα. Έχω δύο-τέσσερα ερωτησούλες όμως. Η πρώτη μερίζα είναι αυτό το οποίο εξηγήθηκε σε σχέση με την ψηφοφορία που είπες για τον εκλογικό νόμο. Εγώ αυτό που θέλω να μάθω είναι το εξής. Σήμερα, σε αυτή τη φάση, οι Λιβανέζοι έχουν λάβει υπόψη τις ε, συστάσεις της ε, αποστολής της οποίας είχε γυθεί ο κύριος Σαλαφράγκα. Επομένως, για πέστε μας. Αυτές οι προτάσεις, οι συστάσεις που κάναμε. Διαμέσου του Ιγνατίου ελήφθησαν υπόψη για τις εκλογές που επίκυνται. Τρίτη ερώτηση. Εάν γίνουν εκλογέ θα γίνουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Γιατί ακόμα στη Συρία συνεχίζει ο πόλεμο φυσικά δεν υπάρχει καμία λύση. γιατί η Χεσμολά ξεχίζει να υποστηρίζει τον τον Άσαντ, και γι' αυτό και έχουμε όλους αυτούς, αυτές τις δεκάδες χιλιάδων και παραπάνω ε, πρόσφυγες που βρίσκονται στο Λίβανο και προέρχονται από τη Συρία. Επομένως, επομένω, ξαπλώνεται παντού αυτή η κατάσταση. Στο βορρά, παντού. Στις πόλεις του Βορείου Λιβάνου τώρα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχοντας επομένως το σενάριο του να μην γίνει αποδεκτός ο κλικός νόμος. Τι έχει μπορεί να πει μας ενδιαφέρει σε σχέση με το τι θα γίνει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την δολοφονία Χαράρη και επομένως και αυτό έρχεται να προσθεθεί σε όλη αυτή την πύρητη δαποδίκη Και επίσης να έρχεται και αυτό να βαρύνει την Χεσμπολά για όλες τις Τρομοκρατικές ενέργειες. Και το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε για αυτή την περιοχή είναι το να έχουμε μια νέα έκρηξη. Ενώ σε αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ε, συγκρατηθεί η κατάσταση. Ε, Διαλέξαν επομένω μέχρι σήμερα επιτυχώ την ε, αποστασιοποίηση από την Συρία, αλλά γι' αυτό σα λέω τι θα κάνουμε, μέχρι πού θα φτάσουμε. Θα γίνουν τα πράγματα σε σχετικά ειρηνική συγκυρία. Και επίσης ελήφθησαν ή όχι υπόψη αυτό το οποίο συνέστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον εκλογικό νόμο. Είναι σημαντικό. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τάνοκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ ήθελα να ρωτήσω ακριβώ σε σχέση με Χεσμολάχ κατά πόσον δηλαδή ε, το κοινοβούλιο έχει κάποια επαφή με τους βουλευτές Χεσμολάχ. Επίσης, ε, αν γίνεται κάποια διάκριση εδώ μεταξύ του, του, του, του, του παρανόμου στρατιωτικού ε, κλάδου της Χεσμολάχ και από την άλλη μεριά του πολιτικού σκέλους, το οποίο κατά πράγματο τρόπο λαμβάνει πόρους της Ένωσης και χρωμητοδοτεί τους, ε, τους τρομοκράτες. Επομένως, ε, ε, πρέπει να ερωτηθεί το Συμβουλίο γιατί να μην ε, να μην αμένει κυρίως την με αυτή οργάνωση που άλλωστε συνδέεται με αυτό που έγινε στη Βάνα που σκοτώθηκαν ε, αθώοι, άμαχοι Ισραηλίνοι. Επίσης, για πετε μας. Ε, τι συζητήθηκε σε σχέση με την ε, Συρία. Τι λέει η πολιτική τάξη για ε, την πτώση του Μπάθ, του Αλάσαντ Άλλωστε πάντοτε θεωρεί το Λίβανος ως ε, η χαμένη πατρίδα για τους Σύρους. Ποτέ δεν έχει την εξαρτησία. Και γι' αυτό και έχουμε την... Ε, ε, τι αυτές τις διόρθινες σχέσεις μεταξύ Βηρητού και Δαμασκού. Και τώρα ο κύριος Πέτριν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ομάδας για τη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από κάποιες εβδομάδες πήγα και εγώ στο Λίβανο και η δική μου εντύπωση είναι ότι το, ο Λίβανος είναι η χωάνη για πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Η πρώτη μου παρατήρηση ε, είναι εξή και αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος κύριος ε, Κύριλοφ. Οτιδήποτε και αν κάνουμε σχετικά με τις ε, διάφορες ομάδες, όλα αυτά θα πρέπει να είναι ειλικρινή. Δηλαδή, να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τα πεπραγμένα. Και εάν οι Αμερικανοί φίλοι μας, αλλά και οι Ισραηλινοί, ε, έχουν αποδείξεις ότι υπάρχουν ε, ε, μέλη της Χεσμολά που δολοφόνησαν Ισραηλινούς, θα πρέπει να μας δοθούν αυτά τα αποδοκτικά στοιχεία και να υπάρξουν συνέπειες για τη Χεσμολά. Βεβαίως και γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η Χεσμολά για την ειρήνη, για τη σταθερότητα στο Λίβανο, αλλά και για την ε, ειρνευτική διαδικασία, αν βέβαια αυτή ξαναρχίσει με το Ισραήλ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τις στενές σχέσεις με τη Συρία και με το Ιράν, ε, παρότι και εκεί αυτή τη στιγμή ε, πάρα πολλά είναι ρευστά. Το θέμα όμως είναι η ειλικρίνεια, η να πούμε και να δούμε ποιος δολοφόνησε τους Ισραηλινούς ε, στη Βουλγαρία. Αυτό συμφέρει εμάς αλλά και τη Βουλγαρία γιατί στο δικό της το έδαφος έγιναν όλα αυτά και η Βουλγαρία πρέπει να ενδιαφέρεται το θέμα να εκλειφθεί ως προτεραιότητα. Το δεύτερο που θέλω να πω και ευχαριστώ θερμά την κυρία Μαρίζα Ματίας ε, που έθιξε το θέμα των προσφύγων. Θέλω να πω λοιπόν το εξή ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον ε, Λίβανο με βοήθεια προς τους ε, πρόσφυγες. Ο κύριο Μάριο Ντάβιτ είπε ότι οι πολλοί πρόσφυγες τελικά βρίσκουν κατάλημα σε φίλους, σε συγγενείς, σε βάρος και αυτό και δεν ισχύει και για όλους. Εάν λοιπόν δεν επιθυμούμε να επιδεινωθεί περαιτέρω η πολιτική κατάσταση στο Λίβανο και ήδη σήμερα υπάρχουν ε, ε ριζοσπαστικές κινήσεις ε, οι οποίες ε, αναπτύσσονται βόρειο-δυτικά. Αν δεν επιθυμούμε να επιδεινωθεί η κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τους ε, πρόσφυγες. Και τελευταία μου παρατήρηση είναι εξή. Εγώ θέλω να σας πω, συναντήθηκα με πάρα πολλούς ε, χριστιανούς και διαπίστωσα προς μεγάλη μου λύπη ότι υπάρχουν, υπάρχει και εκεί διάσταση υπόψεων. Όλοι σμένοι είναι φιλοσύριοι, άλλοι είναι αποστασιοποιημένοι και επικριτικοί απέναντι στη Συρία. Η ε, στάση λοιπόν δεν είναι ενιαία. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να κάνουμε τα πάντα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινοβούλιο για να διατηρήσουμε την επαφή με άτομα όπως με τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σινιώρα, ο οποίος ε, για μένα ε, ήταν ε, ιδιαίτερα αξιόπιστος ε, ως μουσουλμάνος, ως άνθρωπος της ειρήνης. Νομίζω ότι μπορεί να επεραμεινθεί της ειρήνης και νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε με τον κύριο Σινιώρα αλλά και με άλλους σε πολύ καλή επαφή. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι όπως έλεγε η κυρία Ντεκάιζερ, αυτές οι εκλογές έρχονται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κλίμα λόγω των της στην ε, περιοχή και κυρίως όσον αφορά το, το, τον πόλεμο στη Συρία. Είχα την ευκαιρία να είμαι επικεφαλή των δύο εκλογικών αποστολών παρατήρηση στο Λίβανο. Πρώτα-πρώτα είχαμε ε, πολύ διόρθυμε συνθήκε γιατί μόλι ε, είχε προηγηθεί η δολοφονία του κ. Χαρίδη και κατόπιν είχαμε την, τις εκλογές μετά από την απόσυρση του, της Συρίας. Και τότε δεν υπήρχαν ε, ψηφοδέλτια να τα ρίξει κανείς αφού διαλέξει, να τα ρίξει στην ε, κάλπη. Οπότε απλώς είχε κάνει ένα χαρτά και έγραφε τους, ε, τους υποψηφίους που προτιμούσε και έτσι έγιναν οι εκλογές. Επίσης, είχαμε κάποιες αλλαγές πάντως προς το καλύτερο και είχαμε επίση τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίο είχε αναλάβει να τη διεξαγωγή των εκλογών και είχε ζητήσει την ομόνια όλων, όλων των ε, δογμάτων, των θρησκειών μάλλον, σε σχέση με την εκλογική διαδικασία. Και όπω τα γνωρίζετε, συνάδελφοι, ο Λίβανο είναι πολύ ιδιαίτερη χώρα. Και έχουμε τον πρόεδρο που είναι Μαρονίτη, ο πρωθυπουργό είναι Σουνίτη και η Σιήτη είναι ο πρόεδρο τη Βουλή να γίνει τέτοια κατανομία αναθρησκεία. Και το δεύτερο λογικό και αυτό είναι κάπως ιδιότυπο. Και έχουμε κάποιο είδου ποσοστώσει ούτω υπήν, όπω είπε ο κύριο ε, Πέτερινγκ. Ε, Τέλο πάντων, κάποιε ρυθμίσει που δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητέ και προσαρμόσιμε στα, στα όσα γνωρίζουμε. Οπότε, γι' αυτό και είχαμε πάρα πολύ ε, μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το σε μέχρι ποιο βαθμό τα κόμματα και ο στρατό έλαβαν υπόψη, όπω ρωτήθηκε, αυτά τα οποία είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε τελικά να βελτιώσουν το εκλογικό του σύστημα. Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει κάποια ελαττώματα και βέβαια οι δυσκολίε είναι η διορυθμία του συστήματο. Και όπω είχε προτείνει και η Γραμματεία, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συζήτηση για να συντονιστούμε ενώπιση των εκλογών και να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ε, συστάσεις μας. Τι έλαβαν υπόψη. Εμείς για το καλό τους τα είπαμε. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά ε, έχουμε αυτή την επιστολή διαφόρων ε, Αμερικανών ε, μελών του Κογκρέσου σχέση με την κήρυξη εκτός νόμου της Χεσμπολάχ το θέμα είναι περίπλοκο. Είναι και κόμμα πολιτικό και ε, υπάρχει και η, η ένοπλη πλευρά, η ένοπλη, ο ένοπλος κλάδος. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε σχέση με αυτό και πολύ καλά το είπε ο κύριος Σας είπε πώς έχουν τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε. Ο δε θα πρέπει αμήλικτα να διώξει τους ε, ενόχους για τις ε, δημοκρατικές ομάδες και τις ε, δολοφονίες. Πάντως, πρόκειται είναι για κολλητικό κόμμα. Οι βουλευτές εκλέγονται με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Και οποιαδήποτε απόφαση θέσεως εκτός νόμου θα μπορούσε να, να ανατρέψει πάρα πολύ την ισορροπή στη χώρα. Μεγάλη προσοχή εγώ σας συνιστώ. Να το σκεφτείτε πολλές φορές πριν ακολουθήσετε τέτοια, τέτοια λύση. Πάντως, κάτι που είναι πιο σημαντικό κύριε Πρόεδρε είναι η τήρηση του εκλογικού δικαίου, του εκλογικού νόμου, ούτω ώστε μέσα από τι εκλογέ να αναδειχθεί κάποιο κόμμα, να λάβει την ε, κυβέρνηση και να βοηθήσει να επιτευχθεί η εθνική ενότητα στη χώρα. Πολύ για ανάλυση πρέπει να κάνουμε. Και όπως και η κυρία και εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι εδώ την ώρα της ε, εισήγησης. Και να δούμε κατά πόσον θα βοηθήσει ο εκλογικός νόμος για κάποιες ε, δίκαιες, καθαρές εκλογές, ούτως ώστε κάτι να γίνει επί τη βάση των, των ιδιορυθμιών αυτών της χώρας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Ματίας, μήπως θέλετε να σχολιάσετε. Mm. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για όλα σας τα σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τα σχόλια γιατί συμφωνώ με τα περισσότερα. Για τις ερωτήσεις όμως θέλω πρώτα να απαντήσω για το θέμα της Βουλγαρίας, του πύργου, του Μπουργκάς. Αν συζητήθηκε δηλαδή αυτό το θέμα στην αποστολή. Ναι, το συζητήσαμε με τους πολιτικούς και με άλλους εκπροσώπους των Λιβανικών αρχών και θα ήθελα δύο πράγματα να σας πω. Πρώτον, ο Λιβανέζος Πρωθυπουργό μας είπε ότι είναι διατεθειμένος για πλήρη συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές για να βρεθεί ο ένοχος της επίθεσης στον Μπουργκάς. Αυτό το δήλωσε ρητά και μίλησε και για την ανάγκη ολόκληρη διαδικασία και όλα να γίνουν γνωστά και με διαφανή τρόπο η δίκη που θα γίνει πρέπει να γίνει με βάση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και όπως είπε και ο κύριος Σαλαφράγκα πρέπει να επιδειχθεί και ιδέουσα φρόνηση. Αλλά ξανατονίζω ότι ήταν πάρα πολύ πρόθυμες οι αρχές του Λιβάνου να συνεργαστούν και να χορηγηθούν όλα τα στοιχεία. Δεύτερον, στις συζητήσεις μας με τους ηγέτες των διαφόρων κομμάτων και με τους εκπροσώπους των αρχών, ανεξάρτητα από την κομματική θέση του καθενός ή την πολιτική, τον πολιτικό του προσανατολισμό, όλοι χωρίς καμία εξαίρεση ζήτησαν να επιδειχθεί μεγάλη φρόνηση από την Ευρώπη κατά την εξέταση του θέματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κρύψουν ποιος είναι ο ένοχος, όχι. Αλλά μας ζήτησαν να επιδειχθεί φρόνηση και προσοχή. Ακόμη και κόμματα που έχουν, που είναι στην αντιπολίτευση και που είναι κατά του Χεσμπουλά ζήτησαν και αυτά φρόνηση για να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες στο Λίβανο και να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρέμβασης. Απ' τη μία δηλαδή υπάρχει η ευθύνη και από την άλλη οι επιπτώσεις. Και όπως είπε και ο Μάριο Νταβίντ, καλό θα ήταν η Επιτροπή μας να τα συζητήσει. Αυτά δεν έχει νόημα να μην το κάνει. Όλοι οι πολιτικοί πάντως του Λιβάνου εξέφρασαν αυτή τους την ανησυχία και την επιθυμία για φρόνηση για να μην υπάρξει βιασύνη και προχειρότης και για να αποφύγουμε έτσι άχρηστα προβλήματα η έρευνα έχει αρχίσει και θα προχωρήσει απρόσκοπτη. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου μας και εγώ και οι τρεις άλλοι. Δεν πήραμε θέση βέβαια, ακούσαμε απλώς τις τοποθετήσεις των διαφόρων κομμάτων και των εκπροσώπων των αρχών, αλλά δεν τοποθετηθήκαμε. Γιατί η συζήτηση θα γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχω εγώ την απόψή μου, έχει και ο Μάριο τη δική του. Και θα ήθελα να προσθέσω απλώς ότι οι όλοι απέκλεισαν την περίπτωση να δακτυλοδειχτεί αμέσως το Χισμπουλά ως τρομοκρατική υπεύθυνη οργάνωση και ξαναλέω για εκατοστή φορά μαζί της ανφρόνηση γιατί αλλιώς μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και να αμφισβητηθούν, να υπονομευθούν και οι σχέσεις μας. Πάντως η διαδικασία θα είναι διαφανής, αξιόπιστη και θα επιδειχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία. Τα άλλα θέματα τώρα. Η Βερονίκ ο κύριος Σαλαφράγκα έθεσαν το θέμα των συστάσεων της αντιπροσωπείας μας για την ειδική διαδικασία, ε, για την εκλογική εκλογική διαδικασία. Κατανοούμε ότι οι Λιβανέζικες αρχές έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Ένωση, με τα θεσμικά της δηλαδή όργανα, με το Κοινοβούλιο και μας είπαν μάλιστα ότι με την προοπτική των εκλογών πολλοί στο Λίβανο θα θεωρούσαν ευκταία την έλευση μίας αντιπροσωπείας παρατηρητών από την Ένωση. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στις συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε γραπτός. Δηλαδή, υπάρχει το θέμα της συζήτησης του εκλογικού νόμου που είναι εσωτερικό θέμα και αφορά μόνο τον Λίβανο και τους πολίτες του και μόνο εκείνοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν λοιπόν όρια στις συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Οι Λιβανέζικες αρχές λοιπόν και ο λαός θα καθορίσουν τον εκλογικό νόμο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί όπως εκείνοι στη συνεργασία και Πιστεύουμε ότι έχει τεθεί σε σωστές βάσεις ήδη γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ Λιβανέζικων αρχών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τώρα η Συρία. Η κατάσταση στη Συρία επηρεάζει φυσικά και την κατάσταση στο Λίβανο και γι' αυτό οι αρχές του Λιβάνου προσπαθούν να διατηρήσουν την εθνική ενότητα και την εθνική τους κυριαρχία και να μην τοποθετηθούν ως προς τον εμφύλιο ή την κρίση όπως θέλετε στη Συρία. Ένας συνάδελφος είπε ότι υπάρχουν διαφωνίες και μεταξύ των χριστιανών, αλλά τέτοιες διαφωνίες υπάρχουν σε ολόκληρη την Λιβανέζικη κοινωνία. Μερικοί είναι υπέρ του καθεστώτος Άσαντ και άλλοι όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι Λιβανέζικες αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν, το ξαναλέω ακόμη μια φορά, την εθνική κυριαρχία για να μπορέσει να συνεχίσει η εκλογική διαδικασία γιατί όλοι τις θέλουν τις εκλογές. Όσες διαφωνίες και να υπάρχουν μεταξύ κομμάτων και μέσα στην κοινωνία. Οι αρχές πάντως θέλουν πάση θυσία να διατηρήσουν την ενότητα της χώρας και αυτό πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα. Τώρα για το θέμα των προσφύγων. Ο Μάριο μας είπε ορισμένα πράγματα, αλλά είναι φανερό ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρόκειται για πρόσφυγες που γίνονται δεκτοί από οικογένειες και κοινότητες. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο, κατάσταση δύσκολη και απαράδεκτη η αντιπολίτευση προσπαθεί να δημιουργήσει στρατόπεδα προσφύγων όπως ήταν πριν και υπάρχουν ακόμα στρατόπεδα Παλαιστινίων στο Λίβανο. Πρόκειται όμως για ανθρώπους που τους λείπουν τα πάντα και δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Ο ΙΕ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μεγαλύτερος δωρητής να συνεχίσει την βοήθεια για τους πρόσφυγες και να αυξηθεί αν γίνεται γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των προσφύγων. Και προσθέτω ότι η αύξηση του αριθμού των προσφύγων και οι συνθήκες τις οποίες διαβιούν δημιουργούν περισσότερες εντάσεις μέσα στη Λιβανέζικη κοινωνία και αυτό μπορεί να χειροτερέψει πολύ αν δεν υπάρξει στήριξη από τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος. Τέλος λέγω. Θα ήθελα να δηλώσω ρητά ότι στην αντιπροσωπεία αυτή, στην αποστολή αυτή καταλάβαμε πολύ καλά ότι οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Λιβάνου έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια γιατί υπήρξε κλίμα πραγματικής εμπιστοσύνης μεταξύ Λιβανέζικων αρχών και ευρωπαϊκών οργάνων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ενωσιακή αποστολή ή πρεσβεία, αν θέλετε, στο Λίβανο έχει θετικό έργο που πρέπει να συνεχιστεί. Να μην ξεχνάμε το πρόβλημα πάντως των προσφύγων και ιδιαίτερα το πρόβλημα της επίθεσης στη Βουλγαρία. σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές μας. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και σε ένα πενταλεπτάκι πρόκειται να ακούσουμε και κλεισμένον των θυρών τον κύριο Ρούπερτ Τζοϊ που είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας στο Μάροκο. Παρακαλώ, μόνο αυτοί που προβλέπονται να μείνουν στην αίθουσα. Και, που σήμερα σε ο κύριος Τζόι θα έρθει. Chairman, just as a matter of interest, what does... Πρόεδρε, τι εννοείται ακριβώς και κλεισμένων. Ποιοι πρέπει να φύγουν. Ποιοι προβλέπετε να είναι εδώ. Τόσο μικροφόνο ο Πρόεδρος. Όχι, όχι. μένει χωρίς κοινό.